Uh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε. Θα ψηφίσουμε αύριο. Και έχω και μια ανακοίνωση να κάνω. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Ρέιμον Σερνατζότο, ο οποίος φεύγει από την ομάδα του ΕΛΚ και θα